προϊόντων φώκιας. Καταρχήν ο εισηγητής Κριστιαν Σίλβιου Μπουζόη έχει το λόγο. Παρακαλώ έχετε την καλοσύνη κυρίες και κύριοι και εγκαταλείψατε την, εγκαταλείψατε την αίθουσα ε, με ησυχία για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον συνάδελφο. Thank you very much, ε, Mr. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Κοινοβούλιο για τη συνεργασία τους. Χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία τον Ιούνιο υπό τη Λετωνική Προεδρία, η οποία ευθυγράμισε τους κοινοτικούς κανονισμούς με την απόφαση του ΠΟΕ. Το 2009, μέσα στα πλαίσια του βασικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να απαγορεύσει την εμπορία προϊόντων φώκιας, εκτός από τη θύρα των Ινουίτ και άλλων αυτοχθόνων πληθυσμών, η εξαίρεση IC, καθώς και τη θύρα που έχει στόχο την βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μικρής κλίματας και μη κερδοσκοπικού σκοπού, εξαίρεση MRM. Άρα, τα προϊόντα που προέρχονται από τη θύρα της φώκιας δεν βρίσκονται πλέον στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός ε, για την εμπορία προϊόντων φώκιας στην ουσία αμφισβητήθηκε από τον Καναδά και την Νορβηγία στα πλαίσια του ΠΟΕ και στις 18 Ιουνίου 2013 ε, δεν συμφώνησε ο ΠΟΕ με την εξαίρεση MRM. Ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν κρίνει ότι υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δηλαδή 16 μήνες μετά από την έγκριση της έκθεσης και λίγη στις 18 Οκτωβρίου 2015 θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση μόνο 6 Φεβρουαρίου 2015 για την εμπορία προϊόντων φώκιας, ευθυγραμμιζόμενη με την νομοθεσία του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαίρεση MRM. Δεν συμφωνούν όλοι με την απαλήφθη της εξαίρεσης αυτής και θα ήθελα να σας πω ότι τώρα η τελική συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις ε, του ΠΟΕ. Σε σχέση με την εξαίρεση για τους Ινουίτ υπάρχει μια νέα σειρά προϊόντων σύμφωνα με... και σύμφωνα με τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν τα προϊόντα θύρας να ε, μπουν και να εμπορευθούν στην αγορά έτσι ώστε οι Ινουίτ να, να μπορέσουν να έχουν ένα εύλογο εισόδημα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αυτόν αυτοπροσδιορισμό των Ινουίτ και άλλων αυτόχθονων πληθυσμών, διότι θεωρούμε ότι η θύρα της φώκιας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, του πολιτισμού και της ταυτότητας των Ινουίτ, έτσι ώστε να έχουν και εισόδημα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιβιώνουν στις μικρές τους ε, κοινότητες. Μέσα στα πλαίσια ε, του πολιτιστικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αντιπραγματισμού. Πρότεινα λοιπόν ένα νέο άρθρο, το 5α, σε σχέση με τα νέα προϊόντα που θα τεθούν στην ευρωπαϊκή αγορά που είναι απότοκα αυτής της ε, θύρας αλλά που είναι νόμιμα. Τέλος, ε, στο άρθρο 7 ζητήσαμε η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2019 να ε, κάνει έναν απολογισμό για τους νέους κανόνες και την επίπτωσή τους τις επιπτώσεις τους. Ε, προσμένω τις ε, υποδείξεις ε, και τις, τις υποδείξεις σας. Ο Επίτροπος Βέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Σώματος. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Μπουσόη και τους συναδέλφους γιατί τάχιστα δέχτηκαν την πρόταση Επιτροπής έτσι ώστε να αλλάξει ο βασικός κανονισμός για την εμπορία ε, προϊόντων που προέρχονται από τη θύρα της Φώκιας μετά την απόφαση του ΠΟΕ τον Ιούνιο πέρσι. Μέσα στα πλαίσια της απαγόρευσης αυτής, ο ΠΟΕ έκρινε ότι οι εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους Ινουίτ και άλλους αυτόχθονους πληθυσμούς, καθώς και η διαχείριση θαλάσσιων οπόρων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις. Θεωρούμε ότι η επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων οδήγησε σε πολύ καλό αποτέλεσμα και έτσι θα μπορέσουμε να συμβαδίσουμε και να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας ε, με βάση τις υποδείξεις του ΠΟΕ για την εφαρμογή του νέου πλαισίου το οποίο λύγει στις 18 Οκτωβρίου του 2015, τον επόμενο μήνα λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού ε, διευθέτησης ζητημάτων. Χαιρόμαστε διότι μέσα στα πλαίσια του όργανου επίλυσης διαφορών φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να συμμορφωθούμε προς τους κανόνες του ΠΟΕ. Πρόκειται για ένα ε, πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για πολλούς και χαιρόμαστε γιατί βρεθήκαμε, βρήκαμε μία εξισορροπημένη λύση. Μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ήρθαν σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όλα τα κράτη-μέλη και εκείνα που ανησυχούσαν με την πρόταση. Θεωρούμε ότι αυτός ο διάλογος ήταν επικοδομητικός και τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στο τελικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την απαγόρευση με εξαίρεση τους αυτόχθονες πληθυσμούς με βάση τα δεδομένα και του ΠΟΕ και με εξαίρεση βέβαια στη διαχείριση των θαλασσίων πόρων. Θεωρούμε ότι υπάρχει εξισορροπημένη πρόταση έτσι ώστε να τηρήσουμε τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις στον εμπορικό τομέα και να λάβουμε υπόψη και τις ε, κοινότητες τις οποίες αφορούν οι αλλαγές. Λάβαμε υπόψη και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σχέδιο ε, συμμόρφωσης και συμβιβασμού έτσι ώστε να ενημερώσουμε και το κοινό για την απαγόρευση αυτή και τις εξαιρέσεις της. Η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι υποστηρίζουμε την πρόταση σε θέματα ουσίας και ως προς ορισμένα διαδικαστικά σημεία έγιναν ορισμένες αλλαγές και γι' αυτό κάναμε δύο δηλώσεις ε, για τα οριζόντια και θεσμικά ζητήματα τα οποία θα διαβιβαστούν ε, στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως προς τη, ε, το θέμα της έγκρισης του πλαισίου και της χρήσης της διαδικασίας της επιτροπολογίας για το, την τεχνική πτυχή του θέματος. Σας ευχαριστώ. Επόμενος είναι Κρις Forordningen fra 2009 gjorde det ulovligt at sælge selskabs... κανονισμός 1007 του 2009 απαγορεύει την πώληση προϊόντων αποθήρευση φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει καταστροφή για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τους Ινουίτες. Ε, μία από τις ε, εξαιρέσεις ήταν η Ινουίτ ακριβώς και ότι θα έπρεπε να υποστούν τις ε, επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέργησε μελέτη αντικτύπου, αλλά θέλει να εγκρίνει ένα άλλο κείμενο. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο κανονισμός του 2009 ήταν πολύ επιβλαβής για τους Ινουίτ και κατέστρεψαν τις επιχειρήσεις τους. Δεν μπορούν να, να πουλήσουν πλέον τα προϊόντα τους, τα δέρματα. Έχουν τεράστια αποθέματα και έτσι οι κυνηγοί έχουν αποσπαστεί από το παραδοσιακό εμπόριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα διαπραγμάτευση με τον κύριο Μποσόη ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει πλέον υπόψη τα στοιχεία που δεν είχε λάβει υπόψη στην προηγούμενη κατάρτιση της νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βοητσεχόφσκι, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή Γεωργίας αποφαίνεται θετικά επί της έκθεσης. Βεβαίως και θέλουμε περιορισμούς όταν πρόκειται για την εμπορία φωκιών λόγω της βαναυσότητας της θύρας. Θυμάστε τι είχε πει ο Μαχάτμα Γκάντι ότι αξιολογούμε τον πολιτισμό μας με βάση τη μεταχείριση των ζώων από τον πολιτισμό αυτό. Η αγριότητα ε, δεν σημαίνει μόνο αγριότητα σε βάρος των ζώων, αλλά σε βάρος της δικής μας αξιοπρέπειας. Η αγριότητα στα ζώα ε, έχει αρνητικό αντίκτυπο και σε μας. Γι' αυτό είναι θετική η απαγόρευση. Πρέπει όμως να δούμε την ιδιαιτερότητα των γηγενών, των αυτοχθόνων, των Ινουίτς. Κάποιες εξαιρέσεις δηλαδή θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό, το δονίζει η έκθεση και εγώ σαφώς είμαι υπέρ. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ βεβαίως θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπουζόη. Ευχαριστώ για την εφαρμογή των κανόνων ΠΟΕ. Σαφώς η εσωτερική αγορά μας θα λάβει υπόψη του όρους που θέτει ο ΠΟΕ και είμαι ευγνώμων διότι αυτό το καταφέραμε και στην Επιτροπή ε, Προστασίας Καταναλωτών. Το ερώτημα είναι στο μέλλον πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε προστασία των ζώων αφενός αλλά και τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και περιορισμούς. Οι εξαιρέσεις ε, εδώ ε, λαμβάνουν υπόψη την ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Βεβαίως, οι νομικές δυνατότητες που προβλέπονται και επιτρέπονται στα πλαίσια της διαδικασίας του ΠΟΕ διατηρούνται και θα πρέπει να είναι ε, επιτρεπτές ε, για να ε, εγκρίνουμε το κείμενο. Θα πρέπει να, να δούμε, κύριε Επίτροπε, τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα δοθεί στο κείμενο αυτό, αλλά νομίζω ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου είναι επιτυχής. Ε, κυρία Σαλντεμόζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, αυτή τη βδομάδα θα ψηφίσουμε για την ε, τροποποίηση ε, των εξαιρέσεων στο εμπόριο Φώκιας με, στα πλαίσια του ΠΟΕ. Η ομάδα μου συμφωνεί με το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα γιατί το κρίνει θετικά ε, βρίσκει σωστή ισορροπία μεταξύ τριών συνιστοσών και σημαντικών θεμάτων, ε, εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ και των διεθνών δεσμεύσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγόρευση στο εμπόριο φώκιας και υποστήριξη των Ινουίτς των αυτοχθόνων που και συνεχίζουμε να ε, υποστηρίζουμε ε, την ε, οικονομία της σε αυτά τα μικρά πλαίσια για την επιβίωσή τους. Ενημερώνουμε και την κοινή γνώμη και τις αρχές ότι τα προϊόντα φώκια στον Ινουίτσε κυκλοφορούν νόμιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι σημαντικό για την επιβίωση της, αυτο, της κοινότητας αυτής των αυτοχρόνων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό από τη προτινόμενη νομοθεσία. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μπουσόη για την εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ. Επόμενος είναι ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το, την ομάδα του ECR, η, συμβα, η συμβατότητα με τους προδιαγραφέ του πότε είναι το πιο σημαντικό σημείο και σε ό,τι αφορά υποστηρίζουμε την ε, διαγραφή της ε, εξαίρεσης ε, MRR και επίσης να διευκρινίσουμε την εξαίρεση των Inuit. Όχι μόνο να μπορούν να καταναλώνουν οι ίδιοι τις φώκες που θηρεύουν, αλλά να μπορούν να τις πολλούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα στην Γερλανδία, όπου δεν υπάρχει άλλη πηγή εισοδήματος. Επίσης, ε, διατηρήσαμε την αρχική απαγόρευση και τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ECR, ότι διατηρήσαμε την παλιά νομοθεσία. Τέρος, επειδή έχουμε και την καλύτερη νομοθεσία, είναι πιο σημαντικό να, θε, να θέτουμε απαιτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μελετά τις επιπτώσεις, ε, τις επιπτώσεις ιδιαίτερα σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία, προκειμένου να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι για το μέλλον. Άρα υποστηρίζουμε την ε, συμφωνία και πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα καλό βήμα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Κάλλας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η νομοθετική πρόταση αυτή ήθελε, είχε ως σκοπό να υπογραμμίσει τα νομικά δυνατά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την απόφαση του ΠΟΕ. Κάποια πράγματα φαίνεται ότι είναι τελείως αυλαβή, αλλά μπορούν να γίνουν πολύ δύσκολα όταν σε ό,τι αφορά και την πολιτισμική παράδοση της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η πρόταση για την διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, που είναι συμβατή με την απόφαση του ΠΟΕ, δεν έχει ως σκοπό να ξαναξεκινήσει την συζήτηση για την απαγόρευση των προϊόντων φώκια. Θα παραμείνει η απαγόρευση. Η πραγματικότητα είναι ότι στις ε, χώρες της Βορείου Θάλασσης και της Βαλτική υπάρχουν ακόμα ε, άδειε για θύρευση φώκια. Στην Εστονία, για παράδειγμα, υπάρχουν 50 άδειε που χορηγούνται για τέτοιου είδου θύρα. Και ο αριθμό αυτό ε, δεν πρόκειται να αυξηθεί. Το γεγονό ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προϊόντα που θυρεύονται δεν βοηθάει τον κόσμο να συνειδητοποιήσει την αξία των προϊόντων αυτών. Απλά τα αγνοεί. Τονίζω ότι αυτό δεν αφορά λοιπόν την ευημερία των ζώων, αφορά την βιώσιμη χρήση των πόρων. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τις τρέχουσες πρακτικές και να ανακαλύψει με ποιον τρόπο μπορεί και να σεβαστεί την, την, την απαγόρευση, αλλά και να επιτρέψει να συνεχιστούν οι παραδόσεις, γιατί δεν θέλουμε ούτε απώλεια πόρων, ούτε να καταστρέψουμε οικονομίες. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Επόμενη, η κυρία Χάζενκαμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ιστορική η στιγμή που διανύουμε. Επιτέλους, τα συμφέροντα των ζώων ε, λαμβάνονται πλήρως υπόψη και δεν υπρισχύουν τα εμπορικά συμφέροντα. Το κόμμα για τα ζώα είναι ευχαριστημένο με την απόφαση του ΠΟΕ και για να μην παρανοήσετε, αν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο θα έπρεπε τώρα να απαγορευτεί, είναι αυτό τα προϊόντα θύρευσης φώκιας. Γιατί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ε, φώκες, κυρίως ε, νεογνά, μωρά, ούτε τριών μηνών, τα οποία ε, γδέρνονται ζωντανά. Και γιατί? Για να κερδίσουν ε, μόνο χρήματα εμείς με τη γούνα τους. Είναι λοιπόν ένα περιττό προϊόν μόδας, το οποίο κοστίζει τη ζωή με φρικτό τρόπο σε νέο ζώα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη αποφάσισε το 2009 να περιορίσει την εισαγωγή και την, το εμπόριο. Οι δύο εξαιρεσει. δυστυχώς ε, από τις δύο εξαιρέσεις διατηρείται η μία η θύρα από την Ινουίτ. Αλλά αν θέλουμε να διατηρηθεί ο πολιτισμός θα πρέπει ακριβώς να αποτρέψουμε από τους Ινουίτες, να αποτρέψουμε τους Ινουίτες από το να ακολουθούν τέτοιες πρακτικές. Θα πρέπει να καταργηθούν αυτές οι πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλτες, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με μεγάλη αποτελεσματικότητα εργάστηκαν για την έγκριση των τροπολογιών. Το θέμα είναι συγκεκριμένα πολύ σημαντικό και ο κανονισμός για την εμπορία προϊόντων φώκιας και για μας και για την ομάδα μας είναι πολύ σημαντικός διότι ευθύς εξ αρχής ο σκοπός ήταν η προστασία των ζώων. Τα σώμεθα με δραστήριο τρόπο υπέρ αυτής της διαδικασίας. Οι πράσινοι έδωσαν μάχη για αυτό το θέμα. Μετά την απόφαση του ΠΟΕ δημιουργήθηκαν όμως κάποια προβλήματα και συγκεκριμένα ορισμένες πολιτικές ομάδες προσπάθησαν να εντάξουν όσο γίνεται περισσότερες ε, εξαιρέσεις και αυτό θα οδηγούσε σε αποδυνάμωση του κειμένου. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τον στόχο που πάντοτε είχαμε μπροστά μας κατά τις διαπραγματεύσεις. Οι προσπάθειες αποδυνάμωσης αυτές ε, ευτυχώς δεν επέτυχαν και ήδη στην Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, διασκεδάστηκαν αυτές οι προσπάθειες. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και αργότερα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Το πρώτο προβληματικό ήταν η εξαίρεση για τη διαχείριση των θαλασσίων πόρων. Εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ της διαγραφής και εδώ και η Επιτροπή πρέπει να παίξει το ρόλο της διότι πρέπει να γίνει σαφής εκτίμηση και αξιολόγηση για να διαπιστωθεί αν καταστρατηγούνται οι κανόνες ή όχι. Αν ναι, θα πρέπει να αναλυθεί ανάλογη δράση. Ευχαριστώ. Υπάρχει μπλε κάρτα από εσάς, κυρίες Σόλτες. Δέχεστε. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην προστασία των ζώων. Ε, έχουμε την εξαίρεση των Ινουίτ. Στη Βαλτική έχουμε μικρά νησιά όπου η παράδοση ανάγεται σε χιλιάδες χρόνια στη χρήση προϊόντων φώκιας. Ε, δεν... Ε, εμποδίζονται από το να κυνηγούν τη φώκια, να χρησιμοποιούν δίχτυα και εδώ μιλάμε και για εμπορική χρήση των δερμάτων της φώκιας, του δέρματος. Και αν χρησιμοποιηθεί όπλο, τότε μπορεί να χαθού, χαθεί ένα παραδοσιακό επάγγελμα. Κοιτάξτε, ο κανονισμός επέτυχε συμβιβασμό ε, ε, διασφαλίζοντας και το σεβασμό της παράδοσης της ε, δράσης και επιβίωσης των Ινουίτ και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν από τα προϊόντα αυτά της φώκιας. Δηλαδή η θύρα φώκιας μπορεί να συνεχίζεται από τους Ινουίτ. Όμως αν αποδυναμωθεί, πολύ ο ορισμός μπορεί να οδηγήσει σε πολλές εξαιρέσεις, αποδυνάμωση του κειμένου και αυτό θα ήταν κακό για τις φόγες. Η κυρία Πάρκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως κατανοώ και εκτιμώ ότι οι αλλαγές στηρίζονται στις ε, συστάσεις του ΠΟΕ για την προστασία της φώκιας, ανησυχώ πολύ για τον αντίχτυπο που θα έχει αυτό στις κοινότητες των Ινουίτ ε, που θα επηρεαστούν πολύ από τις αλλαγές αυτές. Ε, ανησυχώ διότι δεν υπάρχει εκτίμηση επιπτώσεων πριν από τις ε, τροποποίησεις. Το 2009 όταν για πρώτη φορά ε, προβλέθηκε η εξαίρεση για τους Σινουίτ το Κοινοβούλιο ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος για τους Ινουίτ που για εκατοντάδες χρόνια στηρίζονταν στο κυνήγι της φώκιας για την επιβίωσή τους. Όμως δεν είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσφατα από τη Γρυλανδία τα νούμερα δείχνουν ότι η απαγόρευση επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά τις κοινότητες αυτές. Για να διασφαλίσουμε ε, ότι δεν θα συνεχιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, τις κοινότητες αυτές ε, όπως προστατεύουμε και την καλή κατάσταση των, της φώκιας. Δεν θα πρέπει δηλαδή να θυσιάζονται, να θυσιαστούν τα συμφέροντα του ενός ε, για χάρη των συμφερόντων των άλλων. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ. Η βιωσιμότητα και η σωστή αντιμετώπιση των ε, πόρων των περιβαλλοντικών πόρων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όμως, εν προκειμένου, ε, δεν κινούμεθα σωστά. 12 ε, εκατομμύρια ε, φώκες υπάρχουν ε, στην περιοχή αυτή και 150.000 είναι το, τα θύματα των κυνηγών κατέτος. αυξάνονται τα νούμερα και προφανώς αυξάνονται και τα κέρδη. οι, νουίτ ε, εδώ και χρόνια ε, τις κυνηγούσαν, δεν υπάρχει εναλλακτικό προϊόν και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ε, περιπτώσεις παράνομιου κυνηγιού. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση των φυσικών πόρων. Ε, να φροντίσουμε επίσης ότι η καθαρά ε, εμπορική θύρα δεν θα πρέπει να συνεχίζεται. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη γενικότερη κατάσταση της Βαλτικής και οι εξαιρέσεις να ε, τηρούνται σε συγκεκριμένα όρια. Οι προσπάθειές μας θα πρέπει να αναβαθμιστούν ούτως ώστε οι καταναλωτές στην Ευρώπη να καταλάβουν την ε, διαφορά μεταξύ ε, θύρας για εμπορικούς σκοπούς ε, και θύρας από παραδοσιακές κοινότητες όπως τον Ινουίτ. Σας ευχαριστώ κύριε Ποσπισίλ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κύριο εισηγητή. Ο συμβιβασμός αυτός είναι καλός και πιστεύω ότι η απαγόρευση του εμπορίου σε προϊόντα φώκιας είναι κάτι το ηθικό, κάτι το θετικό που περιορίζει το πόσο υποφέρουν τα ζώα. Βλέπουμε όμως ότι παραμένει μια εξαίρεση. Θα ήθελα να πω από φιλοσοφική, αν θέλετε οπτικής γωνίας ότι αν υπάρχει μία εξαίρεση σε οποιοδήποτε νόμο, αυτό υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες πάντα απαραίτητος. Και ανησυχώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξαίρεση για τους Ινουίτ. Είναι πολύ περίπλοκη, πολύ, πολύ σύνθετη ως εξαίρεση. Έχει πάρα πολλά μικρά τμήματα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να επιτηρείται το κατά πόσον ε, δηλαδή, η εξαίρεση εφαρμόζεται ως προβλέπεται. Αναφέρεται ε, ότι θα πρέπει να είναι μια εξαίρεση για μη εμπορικούς σκοπούς και ότι θα πρέπει να είναι ανθρώπινο το κυνήγι. Αυτό θα το επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων των ζώων και των συμφερόντων της κοινότητας των Ινουίτ. ελπίζω λοιπόν να μην θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το έργο της τελείωσε στην εφαρμογή. Μπλε κάρτα, λέει η Πρόεδρος. Θα απαντήσετε από τον κύριο Όμπερμαϊερ. Θα απαντήσετε στην πλεκάρτα. Ο κύριος Όμπερμαϊερ λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα ότι ο προλαλής σας ανέφερε ότι ανησυχεί για τις εξαιρέσεις που μπορούν πάντα να οδηγήσει σε ζητήματα που δεν τα επιθυμούμε. Δύο Πώς τοποθετείτε σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ε, συντήρησης σε τρόφιμα των αυτόχθονων παραδοσιακών πληθυσμών και κατά δεύτερον θεωρεί επίσης ότι είναι βιώσιμο και ευφυές να καίγονται τα δέρματα των ζώων αυτών. Να πηγαίνουν δηλαδή τελείως άχρηστα. Η απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας, συνάδελφε. Δεν είμαστε εδώ πέρα αντιμέτωποι μεν κατά τον δε. Εγώ ως δικηγόρος, ως νομικός, απλά αναφέρω ότι η εξαίρεση είναι διατυπωμένη με πάρα πολύ περίπλοκο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως καθήκον να παρακολουθεί κατά πόσον εφαρμόζεται ως πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι οι Ινουίτ θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να κυνηγούν φώκες. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο είναι απαραίτητο για την επιβίωση του πληθυσμού, αλλά θα πρέπει να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσον ε, πραγματικά εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Κυρία Γκέπχαρτ τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το 2009 ψηφίσαμε τη γενική απαγόρευση της πώληση προϊόντων και της εμπορευματοποίησης των προϊόντων φώκιας. Ήταν καλό αυτό και θετικό. Αλλά δικαίω προβλέψαμε μία εξαίρεση για τους Ινουίτ. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό αποτελεί βάση επιβίωσης για τον πληθυσμό αυτό, χωρίς την κυνήγη αυτό, χωρίς τα προϊόντα που προκύπτουν από τη θύρα αυτή, πολύ απλά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε απλά να αποφανθούμε ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτή η εξέρεξη ή ότι είναι δύσκολη και περίπλοκη στον έλεγχό της. Όχι. Θα πρέπει να σεβαστούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μια βάση για να επιβιώσουν. Και τότε λοιπόν είχαμε αποφανθεί υπέρ της εξαίρεσης. Η δεύτερη εξαίρεση ήταν λίγο πιο δύσκολη. Ήταν δύσκολη η εξαίρεση. Γιατί η διαχείριση θαλάσσιων πόρων μπορεί να περιλαμβάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Τι μπορεί να κρύβεται λοιπόν πίσω από τη διαχείριση θαλάσσιων πόρων. Είναι θεωρώ θετικό ότι πλέον καταργείται αυτή η εξαίρεση. Εκεί νομίζω ότι είναι θετικό το βήμα που λάβαμε και νομίζω ότι αύριο μπορούμε με ελαφριά την καρδιά να ψηφίσουμε υπέρ του συμβιβασμού γιατί θέτει τι σωστέ προτεραιότητες και επίσης ε, επιτρέπει και μελλοντικό έλεγχο για να δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Ινουίτ γιατί δεν θέλουμε να τους πάρουμε τον τρόπο επιβίωσή τους. Σας ευχαριστώ, κύριε Σφεντερλέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω στη θέση του Προέδρου. Θα ήθελα να σας πω ότι ένα πολύ καλό στοιχείο είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ευημερία των ζώων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια των ε, διεθνών συνθήκων ε, εμπορίας βεβαίως. Μπορούν οι Ινουίτ να συνεχίσουν με την παραδοσιακή τους δραστηριότητα θύρας της φώκιας. Όμως το αρνητικό είναι ότι δεν μπορούμε να ε, ξεχωρίσουμε το, τους δύο αυτούς τύπους θύρας. Ας πούμε στη Σουηδία υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο, όμως το Κοινοβούλιο μας λέει ότι ακόμα και εάν γίνεται θύρα νόμιμη μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης του περιβάλλοντος, ε, παρόλα αυτά μπορούμε να σκοτώνουμε φώκες. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Πράγματι θα θέλαμε να απαγορεύσουμε τη θύρα της φώκιας, αλλά ε, το ζήτημα είναι εκπληκτικό γιατί συνεχίζεται η θύρα της ε, φώκιας και η Επιτροπή το αναγνωρίζει ακόμα και μέσα στα πλαίσια των εξαιρέσεων που υπάρχουν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός ολοένα και αυξάνεται και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε. Δεν είναι σαφές το που βρισκόμαστε και αυτό που εγγράφεται στο νόμο είναι παράλογο. Παρά τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, θα υπήρχαν άλλες δυνατότητες για να επιληθεί το πρόβλημα και η Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να προβούμε στην πλήρη απαγόρευση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την θύρα αυτή η οποία δεν ευσταθεί δεοντολογικά και θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ε, τη θύρα για εμπορικούς και μη λόγους. Αλλά στην ουσία τι κάνουμε. Ε, δεν κάνουμε τίποτα. Ε, προβάλλουμε ημίμετρα. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναγράψουμε τον αγωνισμό εκ του μηδενός. Ο κύριος Νίλσον έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στη Βαλτική. Η εξαίρεση που είχε προβλεφθεί με την απόφαση αυτή καταργείται και αυτό δεν είναι θετικό. Η θύρα της φώκιας στη Βαλτική αυξάνεται σταθερά και αυτό που χρειάζεται είναι μια ισορροπία στο βαλτικό οικοσύστημα. Το πρόβλημα είναι, και το είπα ξανά και ξανά στην Επιτροπή, για να αιτιολογήσω γιατί είμαι κατά της διαγραφής της εξαίρεσης, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίζουμε τους κυνηγούς της φώκιας και αν ακολουθούν τις διαδικασίες που πολλές φορές είναι γραφειοκρατικές. Τώρα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τους σοβαρούς κυνηγού που θέλουν να διατηρηθεί το οικοσύστημα και το, η φώκια, δηλαδή το είδος που κυνηγά. Το πρόβλημα είναι ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε κυνηγού για ένα κυνήγι απαραίτητο. Δηλαδή μπορεί μετά να ε, κληθούν άλλοι να ασχοληθούν ε, με την ε, φώκια. Θα ήταν πολύ άσχημο αν παρενέβαινε, για παράδειγμα, ο στρατός, οι τμήματα των, τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. γιατί έτσι δεν θα μπορούσαμε, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα μπορούσαμε να φροντίσουμε για την προστασία των ζώων όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye, έξι συνάδελφοι ζήτησαν τον λόγο και αν έχουμε χρόνο θα δώσουμε το λόγο σε όλους. Ο κ. Βοντσελίνα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οριστικές αποφάσεις του ειδικού δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, οι δύο ε, εξαιρέσεις αποτελούν αυθαίρετες διακρίσεις. Εμείς θα πρέπει να εγκρίνουμε ε, μια τροπολογία ούτω ώστε ο κανονισμός να συνάδει με τις αποφάσεις του ΠΟΕ. Ε, δεν, στη, στη, στη, στο κυνήγι από τους Ινουίτε δεν ελήφθη η υπόψη η σωστή διαδικασία αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, λανθασμένη προσέγγιση ε, της θύρας ε, για εμπορικούς σκοπούς. Πρέπει λοιπόν να σταθμίσουμε σωστά τις εξαιρέσεις και την καλή κατάσταση των ζώων και να αποφύγουμε την καταχρηστική χρήση αυτών. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί η προστασία των ειδών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της λαθροθυρίας, όπως συμβαίνει με τις φάλαινες αλλά και τις φώκες. Το εμπόριο προϊόντων φώκιας έχει οδηγήσει στην εξολόθρευση του είδους, γι' αυτό και πρέπει να απαγορευτεί. Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας, στον οποίο θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ως μοναδική εξαίρεση την περίπτωση της θύρας που διενεργείται παραδοσιακά στη Γροιλανδία, από την κοινότητα Ινούιτ όμως και εδώ πρέπει να έχουμε αυστηρές προϋποθέσεις πρώτον η θύρα να ασκείται παραδοσιακά από την κοινότητα δεύτερον η θύρα της φώκιας να συμβάλλει στην επιβίωση της κοινότητας των ινουίτ τρίτον να μην διεξάγεται η θύρα για εμπορικούς σκοπούς και τέταρτον τέλος η θύρα να πραγματοποιείται με τρόπο που να μειώνει τον πόνο και την ταλαιπωρία στα θηρευόμενα ζώα. υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική προστασία της φώκιας παγκόσμια ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιβίωση και τον αυτοπροσδιορισμό της κοινότητας των ινούιτ καθώς η θύρα της φώκιας αποτελεί πηγή ζωής για τους κατοίκους αυτής της δυτικής γροιλανδίας και μέρος της πολιτιστικής τους παράδοσης. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ της ε, θύρας της παραδοσιακής ε, θύρας των Ινουίτ και άλλων αυτοχθόνων πληθυσμών και της ε, υπερβολικής θύρευσης ή θύρας που καταλήγει ε, και στο κάψιμο της γούνας της φώκιας χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα ήθελα να σχολιάσω και ένα άλλο πρόβλημα που δεν αναφέρθηκε. Εγώ προέρχομαι από την ε, Κροατία και στα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί χρησιμοποιούμε ε, ελουροειδή, υπάρχουν ε, ε, ελουροειδοί που θυρεύονται και αυτό αφορά ιδιαίτερα την λεπού. Ελπίζω να ληφθούν μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Σεράος Σάντος. Θα ήθελα να πω ότι όταν υπάρχουν δύο Πορτογάλοι ε, θα ε, διαφωνήσουν. Δεν υπάρχει συνένεση σε αυτό το θέμα. Όμως ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανεκτικότητα προς τους άλλους, γιατί τη στιγμή που πρόκειται για μία μορφή αιώνιας φύρας από τους αυτόχθονες για την επιβίωσή τους, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιτρέψουμε. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη ότι ο άνθρωπος είναι σύστημα, είναι μέρος συγγνώμη, ενός οικοσυστήματος, οπότε δικαιολογείται η θύρα, αλλά δεν δικαιολογείται όταν γίνεται για κερδοσκοπικούς ε, σκοπούς και μαζική εκμετάλλευση. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει αυτή η διάκριση. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Φέντερλε. Την ε, ε, δέχεστε κύριε Σάντος. Τη δέχεστε. Εντάξει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση υπέρ των Ινουίτ, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Βορρά, στη Νορβηγία, ε, και στην ε, Σουηδία υπάρχει μία αρκτική παράδοση, δηλαδή από τότε που αποσύρθηκαν οι παγετώνες ε, ή συρρυκνώθηκαν, προωθήθηκε αυτή η μορφή θύρευσης. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή τι μπορείτε να πείτε στην ε, περίπτωση ε, που η φώκια θυρεύεται και μετά ε, γίνεται, καίγεται το δέρμα της. Τι μπορείτε να πείτε για αυτή τη μορφή θύρευσης. Ευχαριστώ πολύ. Από τη δική μου προοπτική, τα ζητήματα θύρας αγρίων ειδών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για αυτόχθονους πληθυσμούς που ε, προαιώνια προέβαιναν σε αυτή τη θύρα και δεν έχουν άλλους οπόρους. Και έτσι θα πρέπει να δράσουμε με βάση αυτή την προαιώνια δηλαδή διαδικασία. Eh, eh, Η ευρωπαϊκή απαγόρευση εμπορικών προϊόντων με έχει μια μεγάλη ιστορία. Το κόμμα μου, το NVA, και η κυρία Μπρέπουλς ήταν ε, στη γέννηση της απαγόρευσης το 2009. Ήταν μια απάντηση που εδώ και καιρό προσμέναν οι πολίτες ε, για να, μην απαγορεύονται, για να απαγορεύονται προϊόντα άγριου εμπορίου, άγρια στήρευσης ε, στην αγορά μας. Η απαγόρευση διάφορες φορές έχει αμφισβητηθεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και είναι σημαντικό το ότι δίνει το πράσινο φως, ο ΠΟΕ γιατί η απαγόρευση πλέον με τις προσαρμογές που γίνονται ε, είναι ακόμα πιο στεναρή. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο λοιπόν να ταπεξέλθει και να έλθει στο ύψος των ε, απαιτήσεων του ΠΟΕ και να μην τις υπονομεύσει. Και η αντιπροσωπεία μας θα υποστηρίξει λοιπόν αύριο αυτή την συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Μία ε, μπλε κάρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται εδώ. Θα ήθελα να πω ότι ασφαλώς υποστηρίζω την αρχή, την αρχή της προστασίας της ευημερίας των ζώων, καθώς και τον ΠΟΕ. Αλλά όσοι μένουν σε μικρά νησιά, στην Εστονία, στην Σουηδία, όπως εκεί που μένω εγώ, διδάσκονται παραδόσεις χιλιάδων ετών. Πάντα υπήρχαν αυτές οι παραδόσεις και τώρα αυτή την παράδοση τη διατηρούν μόνο οι Ινουίτ. Πώς θα εξηγήσουμε στα παιδιά της κοινότητά μας ότι είμαστε περιβολικά μικροί ως κοινότητα για να εισακουστούν οι ανάγκες μας. Στα μουσεία δηλαδή θα μείνουν αυτέ οι παραδόσει των χιλιάδων ετών. Ο Επίτροπο Βέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συμμετασχόντες στη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή τη διαδικασία με τόσο επικοδομητικό τρόπο παρά τις δυσκολίες και τη διάρκεια της συζήτησης. Τα προβλήματα τα θέσατε κι εσείς. Ο νέος κανονισμός θέλει να διασφαλίσει ότι θεμελιώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων που παραδοσιακά ενέχονται στη θύρα της φώκιας δεν θα ε, επηρεαστούν αρνητικά. Η θύρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και της ταυτότητάς τους και είναι πηγή εισοδήματο. Και αυτό, όπως τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές, συμβάλλει στην ε, επιβίωσή τους. Η εξαίρεση για τη διαχείριση θαλάσσιων πόρων δεν είναι κομμάτι του αποτελέσματος γιατί δεν συνάδει με τον ΠΟΕ. Αυτό είναι σαφές. Να είστε βέβαιοι ότι εξετάσαμε ενδελεχώς κάθε πρόταση που υποβλήθηκε. Αλλά δεν είδαμε δυνατότητα διατήρησης της εξαίρεσης χωρίς να ε, διακινδυνεύσουμε κυρώσεις από τον ΠΟΕ λόγω μη συμμόρφωσης συνεχιζόμενης η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα νομοθεσία θα μπορέσει να συμβιβαστεί και να συμμορφωθεί με τον ΠΟΕ και να έχει ένα νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη και θέματα ε, ηθικής που απασχολούν την κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που δίνετε την στήριξή σας στην προτινόμενη νομοθεσία. Ευχαριστώ και τώρα ο εισηγητής. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε για τα καλά σας λόγια. Κατανοώ ότι η συμφωνία που επετεύχθη δεν ικανοποιεί πλήρως κάποιες χώρες της Βαλτικής ε, και κάποιες σκανδιναβικές χώρες η διαφωνή. Όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε διότι τώρα έχουμε νέα κριτήρια για την εξαίρεση των Ινουίτε και τις συμφωνίες για το άρθρο 7 για την πολλή εκθέσεων. Ε, πιστεύω ε, και μετά τις συναντήσεις που είχαμε ε, με εκπροσώπους από την Ιρλανδία και τη Δανία, διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις συναντήσεις με την ίδια την Επιτροπή, ότι η θύρα από τους Ινουίτ και άλλες αυτόχθονες κοινότητες δεν βλάπτει και δεν απειλεί να βλάψει το οικοσύστημα ε, και τους πληθυσμούς της Φώκιας και δεν γίνεται ποτέ για εμπορικούς σκοπούς. Οι Νουίτς ε, κυνηγούν γιατί έτσι ε, συντηρούν την οικογένειά τους και τις μικρές τους κοινότητες. Οι ανάγκες τους ε, για επιβίωση είναι απλές, μετριοπαθείς, ακολουθούν το για εκατοντάδες χρόνια ως κομμάτι της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και σέβονται και εκείνοι οι ίδιοι την καλή κατάσταση των ζώων. Εμείς ε, ε, έχουμε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα και χωρίς την καλή συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να το τηρήσουμε για να φτάσουμε στη συμφωνία, ώστε να έχει χρόνο και η Κομισιόν για να ετοιμάσει όλες τις επόμενες ε, πράξεις που χρειάζονται μέχρι την καταληκτική προθεσμία του Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ και θα περιμένουμε ενδιαφέρον την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,